Ακολουθεί τώρα η συζήτηση για 7 προτάσεις ψηφίσματος για το Ιράν. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντάκτες. Η κυρία Γκόμες. Το Ιράν έχει μια τεράστια ποικιλία, θρησκευτική, γλωσσική κλπ. Έχουμε πολλές θρησκείες, ζωραστρισμός, σουνίτες, ισίτες κλπ. Είναι ε, έχει ένα τεράστιο αριθμό μειονοτήτων, Κούρδους, Άραβες, Αζέρι κλπ. λοιπά που αντιπροσωπεύουν το 50% του πληθυσμού. Έχουμε μια μέση τάξη, μια μεσαία τάξη και πολλού νέου. Είναι περίπλοκη η χώρα και αυτό φοβίζει το καθεστώς που προτιμάει ένα απλό Ιράν που να χαρακτηρίζεται από ένα θρησκευτικό φανατισμό και μια καταπιεσμένη κοινή γνώμη. Αυτό το ψήφισμα περιγράφει τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, σήμερα τη της τακτικής χρήσης της ποινής θανάτου, ακόμα και για παιδιά. Το διαχωρισμό ανδρών και γυναικών, τις ε, γνωστές καταπιέσεις των μειονοτήτων κλπ. Μέσω αυτού του ψηφίσματος στέλνουμε δύο μηνύματα. Πρώτον, η Ευρώπη βλέπει μια ελπίδα στο πρόσωπο ιδιαίτερα των νέων Ιρανών που ελπίζουμε ότι θα πάρουν τη σκητάλη. Και δεύτερον, προς το καθεστώς, το Ιράν ποτέ δεν θα καταφέρει να αναπτύξει το δυναμικό του χρησιμοποιώντας βία και φανατισμό. Δεν θα μπορέσει αν συνεχίσει να καταπιέζει βία το λαό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Η κυρία Σάκη το λόγο συνάδελφοι, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει να αντλεί την ομιμότητά της από την φροντίδα για τις βασικές ανάγκες των πολιτών. Είναι μία από τις βασικές ανάγκες των πολιτών λοιπόν, που πρέπει να ικανοποιήσει. Άμα δεν το ικανοποιήσει αυτό χάνει οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι καταστροφική για το Ιράν και έχει τοξικά αποτελέσματα για τον υπόλοιπο κόσμο και την περιοχή του. Δεν μπορούμε εμεί να είμαστε αδρανοί όταν βλέπουμε άτομα για μικρό αδικήματα να πηγαίνουν στην αγχώνη, γυναίκες να βιάζονται και άτομα τα οποία καταπιέζονται από το ίδιο το καθεστώς τους. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμορρησία για αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε ότι είμαστε μαζί με το λαό του Ιράν όταν ασκεί το δικαίωμά του ελευθερία σκέψης και έκφρασης και ειρηνική διαδήλωση των αισθημάτων του για τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να προασπίσει τα παγκόσμια αυτά ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από τον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τα εμπορικά συμφέροντα. Μόνο όταν το καθεστώ του Ιράν αποκτήσει νομιμοποίηση από του ίδιου του πολίτε του μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο συνομιλητή σε διεθνέ επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σάκε, ο κύριος Κέλλαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση αυτή ο κύριο κελλαν εχει τωρα το λογο ευχαριστω πολυ κυριε προεδρε η κατασταση αυτη βασιζεται σε, στη δράση μιας δικτατορίας η οποία είναι διαβόητη για τον τρόπο με τον οποίο εξαλείφει τους αντιφρονούντες. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά τις εκλογές του Ινίου. Υπάρχουν εκτελέσεις, βιασμοί, βασανιστήρια που έχουν αυξηθεί έκτοτε. Το Ιράν έχει δει το μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά από την Κίνα τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο δεν αντανακλάται στην, ε, στο ψήφισμά μας. Χθες πήγε στην αγχώνη πέντε κρατουμένους στην φυλακή Εδίν, το καθεστώς του Ιράν, μεταξύ των οποίων Σοχέλα Καντήρη, 28 ετών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν απαγχωνιστεί από το καθεστώς Αυτές οι βαρβαρικές λοιπόν ε, εκτελέσεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με εγκλήματα ή υποτιθέμενα εγκλήματα των κρατουμένων. Είναι μια προσπάθεια να ενταθεί η ατμόσφαιρα βίας και τρόμου, ιδίως μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν διεκδικήσει δημοκρατία και έχουν ζητήσει νέες εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρία Κέλαμ, ο κύριος Σταβάρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ανεξάρτητα από την προσέλευση των βουλευτών σε αυτή την αίθουσα, όταν μιλάμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάμε εξ ονόματος των εκατομμύριων ατόμων που έχουν κατέβει στους δρόμους, κινδύνεψαν τη ζωή τους και το προσωπική τους ασφάλεια στο Ιράν για να διαμαρτυρηθούν κατά των νοθευμένων εκλογών στο Ιράν. <clears throat> Τα εκατομμύρια αυτά Ιρανών μέσα και έξω από το Ιράν περιμένουν από εμά κάτι να πράξουμε. Και γι' αυτό το σημείο εκκίνησή μας δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά η αλληλεγγύη και η υποστήριξη προς το δοκιμαζόμενο λαό του Ιράν, τα εκατομμύρια αυτά ανθρώπων που αγωνίζονται για την δημοκρατία και τα θεμελιώδη ανθρωπινά δικαιώματα και οι οποίοι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτό που φυσιολογικά λαμβάνει υπόψη της μια απλή διπλωματική προσέγγιση. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το σημείο κίνησή μα. Είναι γεγονό ότι η δυτική πολιτική πολλέ φορέ ήταν μια πολιτική απλοποιητική, μια πολιτική αφέλεια σε σχέση με το Ιράν. Είναι γεγονό ότι πάρα πολλέ φορέ η Ευρώπη ακολούθησε τι αμερικάνικε πολιτικέ ή άλλε πολιτικέ οι οποίε απεδείχθησαν λαθασμένε. Πολλέ φορέ δεν θέλησαμε να αποδεχτούμε ότι το Ιράν αποτελεί τμήμα είναι μάλλον ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να γίνει αναγνωριστό σαν μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Όπως έλεγε πρόσφατα ένας ιδανός καλλιτέχνης ότι όλα αυτά έχουν γίνει κάτω από την Ιρανική Δημοκρατία. Τώρα πια δεν θέλουμε να έχουμε μια δημοκρατία αν έχει αυτή τη μορφή αυτή η δημοκρατία. Λοιπόν αυτό το κατασταλτικό, καταπιεστικό καθεστώς βασίζεται όλο και περισσότερο στην βία στις νοθευμένες εκλογές και στην γενικευμένη καταστολή. Ο λαός του Ιράν λοιπόν περιμένει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα από το ψήφισμα το οποίο θα, θα εγκρίνουμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Για δυόμιση λεπτά ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι ξέρουμε ποιε είναι οι πολιτικέ και κοινωνικέ καταστάσει στι οποίε βρίσκονται οι πολίτε τη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράκ. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη παρεμβολή τη θρησκεία στι πολιτικέ αποφάσει και ακόμα και στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν ο φόνο του Μπενούτ Σό, του νέου αυτού, ο οποίο καταδικάστηκε παρά το γεγονό ότι την εποχή του αδικήματο το οποίο υποθέτω διέπραξε ήταν ανήλικο. Είναι μία ακόμα περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταστολής κατά των διανομένων, των ε, δημοσιογράφων, των ομοφιλοφίλων και όλων αυτών που αγωνίζονται για την ελευθερία στο Ιράν. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με το καθεστώ του Μαχμούτ Αχμάτι Νετζάντ, ο οποίο ξεκίνησε την προεδρία του με την άρνηση, την επανειλημμένη του ολοκαυτώματο και με την τι απειλέ κατά του κράτου του Ισραήλ. Από το 2005 ο αριθμό των εκτελέσεων στο Ιράν έχει τετραπλασιαστεί και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου άτομα τα οποία είναι ανήλικοι καταδικάζονται σε θάνατο. Επίσης χρησιμοποιείται συστηματικά χρησιμοποιούνται τα βασανιστήρια στις φυλακές και χρησιμοποιούνται μεσαιωνικές μέθοδοι όπως ο λιθοβολισμός και οι ακροτηριασμοί. Αλλά έχει δυσκολία να αντιμετωπίσει το καθεστώ αυτό τι δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων που έχουν βρει το θάρρο να κατεβαίνουν στου δρόμου και να διαμαρτύρονται για τι νοθευμένε εκλογέ. Ο νεαρό Νέντγκα Άγκα Σόλταν σκοτώθηκε όταν δικαι... ή Νέντα Σολτάν ζητούσε το δικαίωμά τη να είναι ελεύθερη σαν γυναίκα και σαν πολίτη και είναι ένα σύμβολο για όλους που αγωνίζονται κατά τη καταστολή. Πώ θα του βοηθήσει η Ευρώπη. Εμεί έχουμε στη διάθεσή μα το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μια άλλη συγκεκριμένη πρόταση είναι να δώσουμε το όνομα τη Νέντα Άγκα Σολτάν σε δρόμου ή σε πλατείε τη χώρα μα. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μονάχα θα είναι μια ανάμνηση τη θυσία της, αλλά θα ήταν και μια μαρτυρία αλληλεγγύης με την Ιρανική αντιπολίτευση και θα δώσει και στους Ευρωπαίους πολίτες μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κατάστασης που επικρατεί στο Ιράν και η οποία είναι πάρα πολύ ζωφερή. Επίσης, θα ήθελα οι εικόνες της Aung San Suu η οποία έχει τις εικόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, να συνοδευτούν αυτές με τις εικόνες της Νέντα Άγκα Σουλτάν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσουμε στον πρόεδρο Αχματιδετσάν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στο πυρηνικό θέμα όταν καταστέλει το λαό το οποίο ζητά περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία και περισσότερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Για ένα λεπτό ο κύριος Στίβενσον τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενώ εμείς καθόμαστε εδώ και κάνουμε μεγαλόστομες δηλώσεις, ε, εκεί κρεμάνε κάθε τόσο ανθρώπους. Χτες κρεμάσαν άλλους πέντε, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα ε, η οποία είχε συγχωρηθεί από τους γονείς του θύματός της, εν πάση περιπτώσει. Εμείς ακολουθούμε μια ε, πολιτική καταπραϊντική εναντίον ε, κατά του, ε, σε σχέση με το καθεστώς ε, προσπαθώντας να, ε, να είμαστε καλοί μαζί τους για να σταματήσουν τις πυρηνικές ε, δοκιμές και την πυρηνική έρευνα. Παρ' όλα αυτά δεν επιτρέπει το καθεστώς ούτε στους ελεγκτές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μπουν στις εγκαταστάσεις τους. Μέχρι πότε θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική κατευνασμού. Χρειάζεται να επιβάλλουμε ε, σκληρά μέτρα. Μόνο αυτά καταλαβαίνουν οι μουλάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λοχμπίντερ. Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας ο πρόεδρος Μπούζεκ Μα είπε ότι η κατάργηση τη θανατικής ποινή είναι βασικό μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό ισχύει για όλε τι περιφερειε του κόσμου, όπου υπάρχει αυτή η απάνθρωπη και ε, φρικτή ποινή. Και μίλησε και για το Ιράν. Σήμερα στο ψήφισμα που έχουμε ενώπιόν μα, γίνεται λόγο για τέσσερι θανατικές καταδίκες Και οι άνθρωποι αυτοί καταδικάστηκαν σε θάνατο διότι υποτίθεται ότι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μετά τις εκλογές. Αλλά ήταν και οι τέσσερις στη φυλακή εκείνη την εποχή. Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις πραγματικά μπορούν να πάνε σε ε, έφεση και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ε, το Ιράν εκτελεί ανηλίκους. Είναι η μόνη χώρα που ε, αυτό το καιρό εξακολουθεί να εκτελεί ανηλίκους. έχει επικυρώσει το Ιράν τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα και τα Πολιτικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και είναι υποχρεωμένο να ε, εγκρίνει νόμο που να απαγορεύει την εκτέλεση ανηλίκων. Υπάρχει ε, λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχη πρόταση και θα πρέπει ε, να καλέσουμε το Ιράν να προχωρήσει στη θέση αυτού του νόμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και τέλος, θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου και να υποκληθώ σε όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες στο Ιράν που ρισκάρουν πάρα πολλά, διακινδυνεύουν, ρίψο κινδυνεύουν, κατεβαίνουν στους δρόμους, έχουν μεγάλη δράση η δραστηριότητα για να ζητήσουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους που τους αναλογούν και βάσει του Ιρανικού Συντάγματος και η αποφασιστικότητά στο το τους, το θάρρος τους ε, αξίζουν επιφύλακτη αλληλεγγύη μας. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Κάστλα. Κύριε Πρόεδρε, χωρίς μικρόφωνο. Στις 2 Οκτωβρίου φέτος η Ιρανική αστυνομία τελευταία στιγμή επέτρεψε κάποιον να πάρει το αεροπλάνο. Ήταν δικηγόρος από το Ολφατάχ Σουλτάνη που έπρεπε να έρθει στην Ιρεμβέργη να του απονείμει ε, ένα βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχε ε, ε, σε ισχύ το διαβατήριό του και δεν τον άφησαν ταξιδέψει. Άφησαν τη σύζυγό του, η οποία διαπίστωσε τα εξή και σωστά και παραθέτω. Λυπάμαι που σε ένα κράτο που θεωρείται κράτο του Θεού εκτελούνται κάποιε πράξει που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Και τελειώνει εδώ η παράθεση έχει ε, μπει ε, σε διάφορε διεθνεί συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έχει κυρώσει και το Ιράν. Και κάθε χώρα ε, εκεί δεσμεύεται να αφήνει οποιοδήποτε πολίτη και δικό τη να ταξιδεύει. Αυτό το παραβιάζει κατάφορα το Ιράκ. Η περίπτωση Σουλτάνη έπρεπε να μπει στο ψήφισμά μας σήμερα και θα σας παρακαλέσω να το υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσενέτσκι. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για να εκφράσω την ανησυχία μας για την κατάσταση στο Ιράν και ιδιαίτερος την ε, κατάσταση των ε, ανθρώπων στο Κάμπα Σραφ, σύμβολο της αντίστασης. Το Ιράν θα πρέπει να καταλάβει ότι το καθεστώς του δεν έχει μέλλον όσο κρατάει την εξουσία με βία. Και θα πρέπει να εφαρμόσει το ψήφισμα της 24 η Απριλίου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει το το Ιράκ να πάψει να μετακινεί ε, βιαίως ε, Ιρανούς πρόσφυγες στο έδαφος του. Είναι ε, καθήκον μας, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε από την, Ευρωπαϊκή Προεδρία και από την Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί περισσότερο στέλνοντα μια μόνιμη ομάδα και ενδεχομένω και μια ειρνευτική δύναμη για να αποφύγουμε περισσότερε βίε ενέργειε εναντίον αυτών των Ιρανών προσφύγων στο Ιράκ και τη βία μετακίνησή του. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπέλντερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τους τελευταίους μήνες έχει ριζικά επιδεινωθεί. Κλασικό παράδειγμα είναι η καταστολή και ο μηχανισμός του Αχμαντίνε Τζάν με οποιαδήποτε μορφή ε, θέλει να ε, στραγγαλίσει από την αρχή οποιαδήποτε μορφή αντιπολίτευσης. Και όποιος δεν είναι στη φρουρά των ε, Ιρανών επαναστατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τα εξή δύο. Πρώτον, μαζί με τους Αμερικανούς θα πρέπει ως δυτικός κόσμος να επικεντρωθούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπει και το ψήφισμα. Και θα πρέπει να καταλάβει η Τεχεράνη ότι αυτές οι παραβιάσεις είναι απαράδεκτες. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν και σοβαρές συνέπειες. Όταν πρόκειται για εθνικά συμφέροντα, κυρίως οικονομικά, έρχονται διάφοροι πραγματιστές ρεαλιστές και σε τελική ανάλυση σου λένε ότι ε, ο Χομεϊνή είχε την ίδια πολιτική και όταν έφτανε το μαχαίρι ε, στο κόκαλο πάντα επιλέγαμε τα εθνικά συμφέροντα στο βωμό της θρησκείας και της ελευθερίας. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και ο Αραβικός κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόρβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και λίγες μέρες μας είχε επισκεφθεί ο κύριος Μπαρόσο και το ρώτησα τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση της, ε, των σχέσεών μας με το Ιράν και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, χώρα αυτή όπου εκατο, εκατοντάδες άνθρωποι όπου εφήγησαν πολλά άτομα αλλά και στην Ουγγαρία εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ε, φυλακιστεί, κρατηθεί και έχουν κρατηθεί χωρίς δικαστική διαδικασία. Μας είπε τότε ο κύριος Μπαρός ότι αυτό ήταν μια εσωτερική υπόθεση της ε, Ουγγαρίας και η Κομισιόν δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πώς αναφερόμαστε σε μια χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θεωρούμε πρέπει να τους πούμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για μια χώρα η οποία είναι πράγματι μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι καταπατώνται τα δικαιώματα των Ούγγρων και πρέπει να λάβουμε μέτρα γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μορφάη. Η κυρία Κόρχολα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράν θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στι διαπραγματεύσει ειρήνευση για τη Μέση Ανατολή. Δυστυχώ αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα τώρα. Γιατί δεν είναι κράτο δικαίου, δεν είναι κράτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχήν πρέπει εμεί να διαφυσβητήσουμε και τα αποτελέσματα των εκλογών που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο όταν ο Αχμάτι Νετζάτ επανεξελέγει και επίση, έκτοτε η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Μετά από το 2005 ο αριθμός των εκτελέσεων είναι τετραπλάσιος από ό,τι στο παρελθόν. Μετά από την Κίνα, το Ιράν είναι η χώρα η οποία εκτελεί περισσότερους από τους πολίτες της. Και επιπλέον, η ελευθερία έκφρασης και τύπου έχει καταπατηθεί. Είναι πάρα πολλοί υγιέτες αντιπολίτευσης οι οποίοι έχουν φυλακιστεί λόγω των πολιτικών ή ακόμα και των θρησκευτικών απόψεών τους. Και μέσα στο ψήφισμά μας ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτούς τους θαραλέους αντιφρονούντες στο, Ισραήλ, στο Ιράν οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν και να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές αρχές και την ελευθερία έκφρασης και ιδίως τις γυναίκες του Ιράν οι οποίες έχουν παίξει ένα κεφαλαιόδη ρόλο στα πλαίσια των, διαδηλώσεων στην Τεχεράνη μετά από τις εκλογές. Ο κ. Φαντάλεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στο Ιράν υπάρχει ένα ακραίο καθεστώς που ακραία ερμηνεύει το Ιράν, το Ισλάμ και το Κοράνι. Όποιος δεν συμμετέχει είναι εκτός νόμου. Είναι μια χώρα που αγχώνει. Ε, σκεφτείτε τους χριστιανούς χριστιανοί που έχουν γίνει μουσουλμάνοι δεν έχουν ε, ε, μάλλον πρώην μουσουλμάνοι που έχουν γίνει χριστιανοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ζήσουν στο Ιράν και απειλούνται ε, με τη θανατική ποινή ούτε διαδηλωτές είδαμε τρεις μήνες τι έγινε μετά τις εκλογές έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μα είναι τελείως απαράδεκτο και τελείως αδιανόητο πώς ένα δικαστήριο ε, καταδικάζει σε θάνατο διαδηλωτέ. Φανταστείτε, ούτε να διαδηλώσει δεν τολμά το Ιράν και ενδυνεύει η ζωή σου. Θα πρέπει ε, να υποστηρίξουμε στεναρά και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους Διαδηλωτές και να αντισταθούμε και στεναρά απέναντι σε αυτό το ομό και βίο καθεστώς του Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Επόμενη κυρία Αντρικέιν. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χειροτερεύει στο Ιράν. Οι αυθαίρετες ε, προεδρικές εκλογές και οι διαμαρτυρίες που επακολούθησαν δημιούργησαν μεγάλη ένταση, πολιτική ένταση στη χώρα. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάτο του καταλόγου των χωρών ε, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Είναι στη θέση 172 από 175 συνολικά. Μόνο η Ερυθρέα, η Νότιο Κορέα και το Τουρκμενιστάν είναι σε χειρότερη κατάσταση. Η γενική κατάσταση του Ιράν είναι από τι χειρότερε στην χώρα. Τα ιστοσελίδε και τα blogs ε, ε, μπλοκάρονται στο ίντερνετ. Η φορή Μπαμπαγιού, θυμάστε, ε, συνελήφθη και η τύχη της αγνοείται. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει μια αποστολή στην Τεχεράνη για να εξετάσει την κατάσταση των που χειροτερεύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και περνάμε στη διαδικασία ο κύριος Χίγκινς. Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τα σχόλια του κυρίου Τσαρνέτσκι ε, το προηγούμενο Ιούλιο έγινε μια επίθεση στον καταφλισμό Αλάσραφ στο Ιράκ. Μόνο ως βαρβαρότητα και αγριότητα μπορεί αυτό να περιγραφεί. Πολλές ε, ε, περιπτώσεις θανάτων και πολλοί τραυματισμοί και σοβαροί. Θα πρέπει να δείτε το βίντεο για να καταλάβετε τι πραγματικά συνέβη. Ο στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις με σαδισμό και όλες το ευχαριστιόντουσαν. 36 συνελήφθησαν, έκαναν απεργία πίνας και τους άφησαν ελεύθερους μετά από διεθνή ε, επιρροή, διεθνή πίεση μετά από 72 ημέρες απεργίας πείνας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόσφυγες. Έχουν δικαίωμα να κοιμηθούν το βράδυ και το πρωί να ξυπνήσουν με ασφάλεια. Και τι χρειαζόμαστε. Δύο πράγματα, όπως είπε ο κ. Τσενέσκη. Πρώτον, ε, μόνιμη ε, παρουσία ε, διεθνή Τη Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, ε, ε, εξασφάλιση και εγγύηση για του ανθρώπου αυτού του πρόσφυγε. Ευχαριστώ κυρία Ντεκεζέ. Okay. Merci. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Euh, trois petits points peut-être pour euh, compléter ce que... Έχω τα εξή σχόλια για να συμπληρώσω του συναδέλφου. Πρώτον, η κυρία Γκόμε νομίζω είπε πω παρόλα τα όσα συμβαίνουν, παρόλα τα, παρόλο το δράμα που ζητώ Ιράν, ε, πιστεύουμε ακόμα, διατηρούμε την πίστη μας στο μέλλον της χώρας αυτής ε, και στη ζωτικότητα της κοινωνίας των πολιτών της. Δεύτερον, δεν έχουμε υπογραμμίσει επαρκώς το γεγονός ότι καταδικάζουμε τις ε, τελευταίες επιθέσεις αυτοκτονίας στον Παλουτσιστάν. Παρόλο ότι ήταν εναντίον των, φρον, των βασταντικών φρόνων, των φρόνων της Επανάστασης, είχαν και θύματα αθώους, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εναντίον τους παρόλα αυτά είμαστε ε, με το μέρος αυτών που αντιστέκονται ε, κατά της ποινής θανάτου ε, ε, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά αλλά και γενικότερα σε οποιοδήποτε άτομο και αν επιβάλλεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντικέζερ. Δίνω το λόγο στον κύριο Πρέντα τώρα. Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να τονίσω ότι εγώ εκφράζω τη βαθύτατη λύση μου, λύπη μου για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν μετά από τις εκλογές του Ιουνίου. Ένα δείγμα αυτής της επιδείνωσης είναι η βία που ασκήθηκε κατά των αντιφρονούντων και η επιθετικότητα της κυβέρνησης. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία έκφρασης η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα στο Ιράν με τις καταδιώξεις ε, με διώξεις κατά των δημοσιογράφων. Ε, μια άλλη μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι οι βασανισμοί και η θανατική ποινή εφαρμόζονται καθημερινά στο Ιράν. Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πρόσφατα ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν ε, καταδικαστεί και, καταδικα... και εκτελεστεί μετά τις εκλογές έχει αυξηθεί σημαντικά. Θέλω να υποστηρίξω επιπλέον την ιδέα να υπάρξει μια αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα βρίσκεται μονίμω στην Τεχεράνη για να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να υποστηρίξει τα δικαιώματα των αγωνιστών για την ελευθερία στο Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέντα. Και τώρα η κυρία Βέρτμαν Κόλ. Βέρτμαν, Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να τα συζητάμε πέμπτη απόγευμα έτσι στο πόδι. Δυστυχώς έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγοι συνάδελφοι. Πριν από ένα μήνα μιλήσαμε για θανάτωση ε, δημοσιογράφων και σήμερα τη Γουινέα, το Ιράν και τη Σιλάκα και την ολέθρια κατάσταση που επικρατεί. Πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν. Ας βρούμε άλλη ώρα να συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα, τα κατεπήγοντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό θα ήταν να μιλάμε και για το θέμα όταν ζητάμε το λόγο στο ΚΑΤΣΙΑΙ, γιατί αφαιρείται χρόνο από τους υπόλοιπους συναδέλφους έτσι. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία του ΚΑΤΣΙΑΙ και δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Όρμπαν. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να διαβιβάσω τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες ε, των θυμάτων ε, για ε, την τρομοκρατική επίθεση στην επαρχία Σιστάν, Μπαλουχιστάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις απανταχού της και επίσης εκφράζει τη θλίψη της και το πένθος της για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανισχύει βαθύτατα για τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν μιλούμε λοιπόν για αυτό το θέμα, σήμερα μιλούμε για εκτελέσεις ανηλίκων, για διακρίσεις εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε διάφορες μειονότητες. Μιλάμε για περιορισμούς και σημαντικούς ε, της ελευθερίας της έκφρασης. Μιλούμε για ε, κακοποίηση ε, ε, κρατουμένων που δεν τη χάνουν δίκαιης και αντικειμενικής δίκης, καταστολή σε μεγάλη κλίμακα ακτιβιστών και διαδηλωτών και αντιφρονούντων και εκπροσώπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει άμεσες επαφές με το Ιράν και εξέφρασε ανοιχτά και ειλικρινά την άποψή της για την εξέλιξη της κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις παγκόσμιες αξίες και αρχές και αισθάνεται υποχρέωση να εκφράσει την άποψή της και να την εκφράζει κάθε φορά που τα θέματα αυτά ε, παραβιάζονται. Δυστυχώς παρά τις ε, δίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται από τις προεδρικές εκλογές και μετά. Ε, εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο του 2009. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ιράν πάρα πολλά άτομα εκτελέστηκαν. Ένα από αυτά τα άτομα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Πρόκειται ένα από τα άτομα τα οποία θανατώθηκε ήταν ανήλικος παρά τις προσπάθειες τις οποίες έκανε ο πρόεδρος. Suntem προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπόρεσε αυτό το τραγικό γεγονός ε, να αποφευθεί. Επίσης, μας απασχολεί τι θα γίνουν 7 θρησκευτικοί ηγέτες Μπαχάη στο Ιράν, που έχουν συλληφθεί εδώ και 17 μήνες έχουν απαγγελθεί πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες ε, εναντίον τους, κατασκοπία, ε, δραστηριότητες παράνομες κατά του κράτους και τα άτομα αυτά πρέπει να σας πω ότι ακόμη δεν ξέρουν με σαφήνεια ποια θα είναι η νομική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Μετά από τις προεδρικές εκλογές συνελήφθησαν εκατοντάδες άτομα τα οποία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Οι δίκες κατά των ατόμων αυτών συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα κατηγορήθηκαν ε, τέσσερα άτομα και τους επιβλήθηκε η θανατική ποινή διότι συμμετείχαν σε αυτές τις ε, διαδηλώσεις. Θα ήθελα συμπερασματικά να σας πω ότι και εμείς έχουμε τις ίδιες ανησυχίες όσον αφορά την πράσινη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις των γεγονότων και κάθε φορά που μπορούμε ζητούμε από τις ε, αρχές του Ιράν να σέβονται τις διεθνείς τους δεσμεύσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κυρίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την Παγκόσμια Διακήρυξη Προσίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Παγκόσμια Σύμβαση. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η περάσπιση τους στο Ιράν είναι στοιχείο κλειδί για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παγιώσει τον πολιτικό διάλογο και να συνεργαστεί στο μέλλον με το Ιράν. Και για να απαντήσω τώρα στο ερώτημα που μου υπευλήθη, πιστεύουμε ότι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι η κατάσταση στη χώρα αυτή, δεν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να πάει στο Ιράν μια πλήρης αντιπροσωπεία του Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Έχουμε έξι ψηφίσματα. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον συνάδελφο Βανόρδεν για ένα λεπτό. Uh,